Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Και πρώτο σημείο στην εμείς διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ραντζέλ για την αλλαγή του καταστατικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό έχει να κάνει και με την έρευνα που έκανε το Κοινοβούλιο, οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και ξέρω ότι ο Πάολο θέλει να μας ενημερώσει για τα πάντα, οπότε θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα απλώς να σας εκθέσω κάποιες απόψεις με επί της ουσίας για το θέμα. Και να σας πω πώς έχουν προχωρήσει οι εργασίες μας από τη σκοπιά του εισηγητή. Ε, η βασική μας δουλειά για το θέμα αυτό θέλει να εντάξει το καταστατικό το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Δημοσιολαβητή στη συνθήκη της Λισαβόνας και να τα συνδυάσει. Όπως ξέρετε, δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις αλλαγές που έχουν απέλθει στη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε βασικός βασικό μας μέλημα είναι να φτάσουμε στις ευρωεκλογέ με ένα καταστατικό που θα είναι πλήρως σύμφωνο με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Ήδη έχω εκθέσει λίγο πολύ και την άποψή μου λέγοντα το αυτό. Διότι δεν πιστεύω πρέπει να αλλάξει επί τη ουσία ιδιαίτερα το καταστατικό του Μεσολαβητή πιστεύω ότι οι βασικές αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή είναι ήπιας μορφής, ούτως ή άλλως. Έχουμε ακούσει απόψεις ότι πρέπει να δοθούν δεσμευτικές εξουσίες στον ε, διαμεσολαβητή, δηλαδή να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις δεσμευτικού υπεχρεωτικού χαρακτήρα. Αυτό θα το θεωρούσα καταστροφικό. Το βασικό μας επίτευγμα στα πολιτικά μας και τα θεσμικά μας συστήματα και με το βασικό σκανδιναβικό μοντέλο αλλά και γενικότερα με το ευρωπαϊκό και τα περισσότερα μοντέλα που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταφέρει να έχουμε μία έναν θεσμό, μία, ένα πρόσωπο που μπορεί να ασκεί μια εξουσία ήπια, σε αντίθεση όμως με την πιο αυστηρή. Δηλαδή οι διαμεσολαβητές καταφέρουν να συλλέγουν πληροφορίες που άλλοι φορείς, άλλα σώματα δεν καταφέρνουν να τα συλλέξουν. Διότι ακριβώ έχουν αυτή την ε, ε, ανεπίσημη, την ήπια προσέγγιση στα πράγματα. Και όσοι μετά είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των αποφάσεων του διαμεσολαβητή, επειδή αυτό το κάνουν οικειοθελώς, ελεύθερα και χωρίς ε, πιθαναγκασμούς, αυτό τελικά έχει θετική... Ε, επίδραση στη λειτουργία του όλου συστήματο. Δεν θέλουμε να γίνει ο διαμεσολαβητή κάτι σαν εισαγγελέα ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν καταστροφικό. Είναι πολύ χρήσιμο θεσμικό πρόσωπο και λειτουργήμα. Βέβαια δεν έχω ακόμη διαβάσει την έρευνα, αλλά βλέπω να υπάρχουν ε, στον τίτλο ε, και το δυναμικό και τα χαρακτηριστικά του ρόλου του διαμεσολαβητή. Αυτό το δυναμικό λοιπόν είναι ένα θέμα και θα ήταν καλό να σεβαστούμε αυτούς τους βασικούς άξονες λειτουργίας του διαμεσολαβητή, τα θεμέλια του λειτουργήματος. Νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το στόχο μας και εξ όσων γνωρίζω υπάρχει αυτή είναι μάλλον η άποψη και της διαμεσολαβήτριας αυτή τη στιγμή δεν θέλει ουσιαστική αλλαγή στο ρόλο της, στο καταστατικό της. Βεβαίως κάποιες βελτιώσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επιπλέον, επιτρέψτε μου μερικές τελευταίες παρατηρήσεις στα πλαίσια αυτής της βασικής μου εισήγηση για την δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε εδώ. Νομίζω ότι η προσέγγιση όλων μας δεν έχει δείξει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Μιλάμε για ένα θεσμό ανεξάρτητο, αμερόληπτο, ουδέτερο εξορισμού. Καλό είναι λοιπόν αυτό το καταστατικό να εγκριθεί ευρέως από όλου με μια μεγάλη πλειοψηφία και να σας πω ότι βρίσκω πολύ σημαντικό να μην αρχίσουμε τους ορισμούς της κακοδιαχείρισης, να έχουμε ένα θετικό ορισμό ε, και να είναι ευέλικτη, να είναι μάλλον λίγο πιο γενικόλογη όλη η έννοια. Η κακή διοικητική συμπεριφορά μπορεί να είναι και δημιουργική. Το να είναι κανείς εφάνταστος δεν είναι κακό. Να μην προσπαθήσουμε λοιπόν να περιοριστούμε, να περιορίσουμε τους αυτούς μας με έναν αυστηρό ορισμό. Ξέρουμε τις έννοιες, ξέρουμε τα βασικά ζητήματα, ξέρουμε το τι συμβαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μία έννοια αρκετά χαλαρή. Αυτές θα είναι οι βασικές γραμμές ε, που θα ακολουθήσω στη σκέψη μου, οι αδρές γραμμές για να συνταχθεί η έκθεση και να προτείνουμε την αλλαγή στο καταστατικό. Βασικός μας στόχος είναι όλες οι λεπτομέρειες της διατάξης, της ρυθμίσης, απλώς να συνάδουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν κοιτάμε να επινοήσουμε κάτι καινούριο ή να επαναπροσδιορίσουμε όλο το λειτουργήμα. Επεναντίας θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτρέψουμε στον διαμεσολαβητή να λειτουργεί ανεμπόδιστα και στην επόμενη θητεία με το κύρος και τη βαρύτητα που αναγνωρίζουμε ούτως ή άλλως. Αυτός θα είναι ο βασικός μας σκοπός. Just... Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να σας πω, Πάολου, ότι και εγώ πιστεύω ότι η ήπια εξουσία μπορεί να είναι αποτελεσματική, εάν βεβαίως λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο, ένα τοπίο που επιτρέπει την ε, καλή της λειτουργία. Δεν είναι αυτονόητο. Ο λόγος τώρα στην κυρία Κοτανίδη, η οποία εκπροσωπεί το Κέντρο Μελετών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση σας σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε αυτή την ε, δημοσίευσή μας ε, και η παρουσίαση δική μου σήμερα ακολουθεί ακριβώς ε, την ε, δομή αυτής της ε, δημοσίευσης και αναφέρεται ακριβώς στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή και κάποιες σκέψεις σε σχέση με το ρόλο του και το δυναμικό του. Αναλύσαμε λοιπόν το ρόλο του μέσα στην θεσμική δομή και αναλύσαμε το τι ακριβώς κάνει και μάλιστα το αξιολογήσαμε και ε, το ποσοστό συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων με τις συστάσεις του Μεσολαβητή και από εκεί και μετά αναφερόμαστε και στις δυνητικές βελτιώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επέλθουν σε ό,τι αφορά τις σημερινές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή. Ε, κάποιες ε, μεγαλύτερες κλίμακας σε κάποιες μικρότερες κλίμακας. Ποιος όμως ακριβώς είναι ο διαμεσολαβητής. Έχω φέρει μαζί μου κάποιες διαφάνειες στην παρουσίασή μου, αλλά πρέπει να επιτύχω να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιος είναι ο διαμεσολαβητής. Δεν πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο με βάση το άρθρο 13 της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για ε, ένα, όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αποτελεί ούτε δικαστή, ούτε νομοθέτη, ούτε διοικητικό όργανο. Ωστόσο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτός είναι να ε, ασκεί εποπτεία στη διοίκηση. Δηλαδή η συνθήκη αναθέτει στον ε, διαμεσολαβητή να αποκαλύπτει ε, περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ε, και αυτό κατοχυρώνεται και μέσα στο άρθρο 228 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς σε αυτό το πλαίσιο ο διαμεσολαβητής έχει ένα διπλό ρόλο τον, του να αντιδρά σε παράπονα και από την άλλη πλευρά του να αναλαμβάνει ο ίδιο την πρωτοβουλία. Δηλαδή, λαμβάνει παράπονα, για παράδειγμα, από πολίτε, από οποιοδήποτε άτομο το οποίο διαμένει παράνομα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα παράπονα, αυτές οι αναφορές μπορούν να αφορούν ζητήματα κακοδιαχείρισης, την οποία θα αναλύσω και λίγο αργότερα. Και από εκεί και μετά ο διαμεσολαβητή με βάση το άρθρο 228 και με βάση και το καταστατικό του και τι εφαρμοστικέ διατάξει, οι οποίες εξηγούν ακριβώς το πώς ακριβώς ασκεί τα καθήκοντά του, ο διαμεσολαβητή έχει τη δυνατότητα να εκινεί με δική του πρωτοβουλία ε, Κάποιε έρευνε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να είναι ανεξάρτητος. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα εξωτερικό ερέθισμα, αν θέλετε, ένα εναρτήριο λάκτισμα, αν θέλετε, ε, έξωθεν. Μπορεί ο ίδιος να αναλάβει την πρωτοβουλία ο διαμεσολαβητής και με βάση την εκάστοτε κατάσταση, με βάση τα ζητήματα τα οποία θεωρεί σοβαρά, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Με βάση τη συγκεκριμένη χρονική και, αν θέλετε, ιστορική συγκυρία. και επίσης με βάση μια ανάλυση που έχει γίνει μπορεί, ε, αναλαμβάνει και ένα διαμοσολαβητικό ρόλο αλλά και έναν επιμορφωτικό ρόλο. Και, αυτός, ε, και αυτοί οι ρόλοι σχετίζονται ακριβώς με τις έρευνες, με δική του πρωτοβουλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι εξουσίες του, καταρχήν ε, μπορεί να επιτύχει μια ε, λύση φιλική, δηλαδή ενό φιλικού διακανονισμού. Ε, και εδώ ε, καλύτερα να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θέλει να επιτύχει το θεσμικό όργανο και εκείνο που αφορά στο παράπονο, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, η προσφυγή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Για, για παράδειγμα, ε, σε, σε αυτή την περίπτωση ζητείται η πρόσβαση στο σύνολο του εγγράφου, το οποίο όμω ωστόσο δεν θα ήθελε να δημοσιεύσει το θεσμικό όργανο και σε αυτή την περίπτωση προσπαθεί να ε, ωφελήσει και τι δύο πλευρέ ο διαμεσολαβητή, ε, για να βρει δηλαδή με κοινό αποδεκτή λύση. Από εκεί και μετά, ε, σε ορισμένε περιπτώσει μια έρευνα, δηλαδή εκεί όπου πραγματικά διαπιστώνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένδειξη κάκο διαχείριση, προβαίνει σε μια σύσταση, δίνει τρει μήνε σε ένα θεσμικό όργανο για να απαντήσει και από εκεί και μετά μπορεί να ε, προβεί σε μια απόφαση, δηλαδή ότι δεν υπήρξε κακοδιαχείριση ή ότι υπήρξε κακοδιαχείριση. Με βάση λοιπόν αυτό το πόρισμα σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μη κακοδιαχείριση μπορεί να ασκήσει αυτό τον επιμορφωτικό του εντό εισαγωγικών ρόλο. Δηλαδή μπορεί να προβεί σε συστάσει. Μπορεί να πει έτσι πολύ χονδρικά ότι το σύστημα λειτουργεί καλά αλλά μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Και από εκεί και μετά αναφέρθηκα και στις ερευνές πρωτοβουλία του ίδιου του διαμεσολαβητή. Και αυτό είπαμε ότι αποτελεί μια ευρύτερη εξουσία η οποία έχει ε, δοθεί στον ε, διαμεσολαβητή. Δηλαδή όπου εκείνο θεωρεί μπορεί ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία να ε, ξεκινά μια έρευνα. Οι αποφάσει τώρα που λαμβάνει ο διαμεσολαβητή δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα δεσμευτικό δηλαδή εννοείται για το θεσμικό όργανο στο οποίο απευθύνονται. Άρα λοιπόν ένα είδο soft power, δηλαδή πρόκειται για συστάσεις. Συστάσεις με στόχο ακριβώς να πείσουν το θεσμικό όργανο να αλλάξει την προσέγγιση του σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να παρισφέρουν στην ε, άσκηση ε, της δικαιοδοσίας από την πλευρά του δικαστηρίου και επίσης δεν μπορούν να παρισφέρουν στις δραστηριότητες ενός κράτους μέλους. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις του διαμεσολαβητή ε, έχουν ένα σαφή περιορισμό, δηλαδή αναφέρονται στα θεσμικό όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ όταν αναφέρομαι στα θεσμικά όργανα περιλαμβάνω και τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς και τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ε, τι είναι ο ελέφαντας όπως λέμε στο δωμάτιο, δηλαδή κάτι το που είναι το, το βασικό στοιχείο εδώ που μας αφορά, είναι αυτό το ζήτημα της κακοδιαχείρισης το οποίο διέρχονται ο διαμεσολαβητής. Ε, νομίζω πως ε, έχουμε φτάσει πλέον σε έναν ε, κοινό αποδεκτό ορισμό. Διάφοροι διαμεσολαβητέ στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει να βρουν μια κοινό αποδεκτή έννοια, ένα σωστό ορισμό, αλλά ο, ευρύτερα αποδεκτό είναι εκείνο ε, που τελικά δόθηκε από τον κύριο Σόντερμα που ήταν ο πρώτο ε, διαμεσολαβητή το 1997 και όρισε την κακοδιαχείριση ω την περίπτωση όπου ένα οργανισμό δεν ε, δράει σύμφωνα με μια αρχή η οποία είναι δεσμευτική για αυτό. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να, δεν υποχρεωτικά για κάτι το οποίο ε, αναφέρεται κάπου κατοχυρωμένα σε μια συνθήκη, αλλά για μια ευρύτερη αρχή, σιωπηρή. Γιατί όπως έχει πει και ο κύριος ε, ε Διαμαντούρος, προηγούμενος δηλαδή διαμεσολαβητής, ότι υπάρχουν και όλες εκείνες οι περιπτώσεις μια κρίζα ζώνη, για παράδειγμα, σε νομικό επίπεδο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι πολύ συγκεκριμένε αρχέ. Και εδώ, για παράδειγμα, περιλαμβάνεται η έλλειψη ευγένεια, η έλλειψη μέσα απάντηση από την πλευρά ενό διοικητικού οργάνου, η έλλειψη διαφάνεια. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ευρύτερο ορισμό τη νομιμότητα στην οποία αναφέρεται η κακό διαχείριση. Ε, Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπετε ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια να καταγράψουμε τις δραστηριότητες, τη δράση γενικότερα του διαμεσολαβητή και τις επιδόσεις του. Αλλά εδώ ε, αναφέρουμε τους κύριους τομείς, του οποίους αναλαμβάνει η δράση ο διαμεσολαβητής και βλέπετε πως ε, ε, τα πρώτα χρόνια έως το 2015 αφορούν σε μία φορά από διαφορετικούς ε, ε, τομείς της έκθεσης του διαμεσολαβητή. Δηλαδή εδώ βλέπουμε για τα έτη 2009 έως 2015 όχι καλύπτονται. Ενώ τα έτη 2016 έως 2017 ακολουθούν μια διαφορετική κατηγοριοποίηση και δεν εξαρτάται αυτό από εμά. Ο ίδιος ο διαμεσολαβητής άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητες του. Πάντως βλέποντας σε πιο γενικές γραμμές ο βασικός κλάδος αν θέλετε στον οποίο εστιάζει η δουλειά του διαμεσολαβητή είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση δηλαδή σε έγγραφα και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος τομέας ή ο δεύτερος σημαντικότερος τομέας ε, σε ό,τι αφορά το ποσοστό των εργασιών του διαμεσολαβητή είναι η παρακολούθηση των εργασιών της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες σε παραβάση. Και εδώ να πούμε ότι ε, ο διαμεσολαβητής δεν αξιολογεί ε, την ίδια την, την ουσία δηλαδή της υπόθεσης, απλώς διασφαλίζει το ότι η Επιτροπή ασκεί την, ε, τα, τις εξουσίες που έχει στη διακριτική ευχέρεια με το σωστό τρόπο, δηλαδή με βάση έναν συνεκτικό τρόπο, χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις, ε, προστατεύοντας το δικαίωμα προσφύγης και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπε τώρα κατηγορίες, ή τομεί αν θέλετε δραστηριότητας, αφορούν ε, τον θεσμικό ρόλο των οργάνων, και εδώ μιλάμε δηλαδή για μια πολύ ευρεία κατηγορία σε ό,τι αφορά τον θεσμικό ρόλο, στην οποία εμπίπτουν μεταξύ άλλων και όλες οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το γλωσσικό καθεστώς, για παράδειγμα, συγκεκριμένων εγγράφων και ούτω καθεξής. Μιλάμε δηλαδή για μια ιδιαίτερα ετερογενή κατηγορία, η οποία είναι δύσκολο έτσι να οριοθετηθεί πολύ συγκεκριμένα. Μετά έχουμε μια ακόμα κατηγορία που είναι το καταστατικό προσωπικού των οργανισμών. Και εδώ στις αιτήσεις εκθέσεις περιλαμβάνονται στην αλόγω δηλαδή κατηγορία και τα ζητήματα ε, δεοντολογίας και τώρα σύγκρουση συμφερόντων. Και από το 2016 έχουμε μια νέα κατηγορία εδώ, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο για παράδειγμα προαγωγές, αλλά και περαιτέρω ζητήματα ε, πιο ευαίσθητα. Από εκεί και μετά έχουμε και τα, ε, την επόμενη κατηγορία των ε, δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων, δηλαδή όπου, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ε, του εκείνου που προβαίνει στο διαγωνισμό σε ό,τι αφορά για παράδειγμα καθυστερούμενες ε, πληρωμές ε, και ούτω καθεξής. Περνάω στην επόμενη διαφάνεια. Θα ήθελα να σας κάνω μία παρουσίαση σε ό,τι αφορά κάποια βασικά νούμερα. Ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, οπότε εκείνο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι η δραστηριότητα στο επίπεδο τη ίδια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο διαμεσολαβητή και γι' αυτό προετοιμάσα αυτή τη διαφάνεια. Ε, έχουμε δύο διαφορετικά είδη περιπτώσεων όπου από τη μία πλευρά ο διαμεσολαβητη θεωρεί πως ένα ε, ζήτημα είναι ενδιαφέρον και αποστέλει ένα δικό του ερωτηματολόγιο στο εν λόγω θεσμικό όργανο, στον εν λόγω οργανισμό και προβαίνει στα δικά του πορίσματα ή και έχουμε μια δεύτερη κατηγορία εκεί όπου αποφασίζει ο διαμεσολαβητής να διερευνήσει περαιτέρω μια προσφυγή η οποία διαμεσολαβητη να διερευνησει περαιτερω μια προσφυγη η οποια ωστοσο δεν είναι επίσημα παραδεκτή γιατί πρόκειται για παράδειγμα για ένα, μια προσφυγή η οποία δεν εμπίπτει μέσα στο πεδίο αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση ο διαμεσολαβητή μπορεί να αποφασίσει ότι θα προβεί σε μια έρευνα με δική του πρωτοβουλία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει το, ε, την ελόγω προσφυγή ως ε, μη υπαρκτή. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο διαφορετικές ε, περιπτώσεις και έχουμε το ε, κίτρινο από τη μία, την κίτρινη ε, στήλη από τη μία, λέει ο μιλήτρια, και ε, την ε, μπλε. Και έχουμε λοιπόν Είχαμε μια περίοδο του 2011 μια ε, μεγάλη αύξηση γιατί ο κύριος ε, Διαμαντούρος τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ε, τέτοια προσπάθεια σε ό,τι αφορά δηλαδή, την διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων και βλέπετε ότι λειτουργήσε. Έγιναν δηλαδή πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τους, τις διάφορες υπηρεσίες ενώ οι, αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν είναι δεύτερες μετά από την Επιτροπή που λαμβάνουν αυτό τον αριθμό ε, των, ερευνών. Ε, αλλά βλέπουμε πως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ε, σχετική μείωση. Ε, αλλά εδώ δεν μιλάμε για απόλυτους αριθμούς, βέβαια μιλάμε για ποσοστά. Όμως τα ζητήματα τα οποία διαρευνούνται είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου, για παράδειγμα ζητήματα ε, δεοντολογίας, ανάληψης διαφορετικών καθετών, καθηκόντων, ε, όπως αυτό ονομάζεται revolving doors και ούτω καθεξής. Επόμενη διαφάνεια τώρα. Εδώ βλέπετε ότι εγώ έχοντας διαβάσει εκτεταμένη βιβλιογραφία σε σχέση με τον διαμεσολαβητή συμπεραίνω ότι πραγματικά πρόκειται για ένα επιτυχημένο θεσμικό οργάνο. Δηλαδή η συμμόρφωση με τις συστάσεις του είναι ε, πολύ εκτεταμένη. Και εδώ μπορείτε να δείτε για παράδειγμα τη ε, γραμμή, δηλαδή την συνολική συμμόρφωση. Δηλαδή, όχι ε, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις τις οποίες έχει ε, πράγματι διαπιστωθεί μια κακό διαχείριση, αλλά και συστάσεις όπου δεν έχει διαπιστωθεί. Και ο μέσος όρος εδώ της συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλός, ε, δηλαδή το ποσοστό είναι πάνω από 80% και βέβαια είναι ένα καλό ποσοστό γιατί αν ήταν 100% θα σήμαινε ότι δεν είναι αρκετά τολμηρό αν θέλω το διαμεσολαβητή στις συστάσεις ε, που κάνει. Ε, αν πάντως ρίξουμε μια πιο σεκτική μάτια θα διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό συμμόρφωσης με τι συστάσεις, τι περιπτώσεις εκείνες όπου ο διαμεσολαβητής δεν έχει διαπιστώσει κάποια διαχείριση και απλώς προβαίνει σε μία σύσταση, είναι πολύ υψηλό εδώ το ποσοστό, δηλαδή 98%. Αυτή είναι η κόκκινη δηλαδή γραμμή. Εάν ωστόσο ρίξουμε μια, μια ματιά στην κίτρινη, μάλλον πορτοκαλί, ε, γραμμή εδώ, ε, σε ό,τι αφορά τη συστάση όπου υπάρχει ε, διαπίστωση κακοδιαχείριση, βλέπουμε υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωση και μάλιστα με μια ε, μείωση σε 41% το 2015. Αλλά γενικότερα το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό. Και για να κλείσω τώρα εδώ, γιατί αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια που θα εξετάσω, αφού δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας, να σας πω πως ε, το δυναμικό του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή είναι το εξή. Η εντολή του διαμεσολαβητή είναι ενδιαφέρουσα και επίσης είναι ευέλικτη. Δηλαδή, έχουν εκφραστεί απόψει για τον υπέρ του να αναλάβει περισσότερε εξουσίε ο διαμεσολαβητή. Και αυτό έχει υποθεί και από τον ίδιο τον διαμεσολαβητή. Για παράδειγμα, στο παρελθόν ο κύριο Διαμαντούρο είχε αξιώσει ε, πιο ισχυρέ εξουσίε, πιο διευρυμένε εξουσίε σε ό,τι αφορά ε, ε, τέτοιου είδου έρευνε από πλευρά του διαμεσολαβητή και αποφασίστηκε ότι πράγματι θα δοθούν αυτέ. Βέβαια τότε δεν ε, πρόκειται για μια κραυγή βοήθεια από την πλευρά του διαμεσολαβητή, πράγμα βέβαια το οποίο μπορεί να είχε γίνει ανεπίσημα. πάντω. Ε, όσοι από εσά έχετε την υπομονή να διαβάσετε τη μελέτη σας, ε, τη μελέτη μας, θα διαπιστώσετε ότι κάνουμε δύο βασικές συστάσεις. Καταρχήν, να είναι λιγότερο Ε, τις δυτικές προτάσεις, ε, οι συστάσεις που κάνει ο Μεσολαβητής δηλαδή θα μπορούσαν να βασίζονται ε, για παράδειγμα σε βέλτιστες πρακτικέ, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιούνται στο εργαλείο. Και ένα δεύτερο μια δεύτερη δέσμη αλλαγών, θέλετε, που, έχουν πιο, που μεταβάλλουν πιο πολύ το καταστατικό και τη συνθήκη και θα μπορούσαν να έχουν περισσότερο ε, αντίκτυπο στον νερό του διαμεσολαβητή είναι αυτά που θα σας, σας αναφέρω σε λίγο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία, όταν ε, υπάρχει ένα διοικητικό όργανο το οποίο δεν ε, προσαρμόζεται στη σύσταση του διαμεσολαβητή, η έσχατη λύση που έχει στη διάθεσή του ο διαμεσολαβητής είναι να θέσει αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η Επιτροπή ΠΕΤΗ λοιπόν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό και να το παρουσιάσει στην Ολομέλεια. Και βέβαια με βάση αυτή την, τη, σύσταση μπορεί να εμ, συντάξει για να υιοθετήσει ένα ε, ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια αυτή η δυνατότητα δεν αξιοποιείται συχνά. Και ο κύριο Διαμαντούρο είχε πει ότι δεν θα ήθελε να αξιοποιήσει συχνά αυτή τη δυνατότητα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ήδη επιφορτισμένο με πάρα πολλά και δεν θέλω να αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα για οποιοδήποτε είδο κακοδιαχείρισης. Πρόκειται δηλαδή για μια περίπτωση εδώ όπου ε, ο διαμεσολαβητής συχνά δεν αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα της ειδική έκθεσης του Special Report. Ωστόσο, ε, αυτό που έχει κάνει ο διαμεσολαβητής στο παρελθόν είναι ότι θίγει αυτό το ζήτημα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, κάτι το οποίο δεν απαγορεύει το καταστατικό και απλώς αποτελεί μια συνήθεια πρακτική διαμεσολαβητή. Και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει ε, προκύψει στο παρελθόν είναι η αναφορά ε, του, αυτού του ζητήματος ε, του δικτύου των διαμεσολαβητών ε, γιατί βέβαια αυτό το δίκτυο αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τους εθνικούς διαμεσολαβητές γιατί βέβαια ο Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητής δεν έχει αρμοδιότητα για τα κράτη-μέλη οι εθνικοί διαμεσολαβητές έχουν αρμοδιότητα άρα λοιπόν συχνά αυτή η ανάθεση γίνεται στι εθνικέ αρχέ σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που με τη σειρά του βέβαια μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίτυπο σε ό,τι αφορά την αλλαγή τη νομοθεσία γενικότερα. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδου ε, δράσει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά αναφορέ που γίνονται απέναντι στου εθνικού διαμεσολαβητέ ή και στον Ευρωπαίο, είναι κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο καταστατικό και θα μπορούσε ενδεχομένω να περιληφθεί. Κάτι ακόμα το οποίο με απασχόλησε λίγο είναι η ποιοτική αξιολόγηση ε, τη. Ε, ε, συμμόρφωση, γιατί έχουμε πολλούς αριθμούς ε, στη διάθεσή μα, αλλά για παράδειγμα δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί, όπω είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, υπάρχει χαμηλό ποσοστό σε ορισμένε περιπτώσει συμμόρφωση με τι συστάσει. Για παράδειγμα, αυτή η κίτρινη γραμμή, η πορτοκαλή γραμμή στην προηγούμενη διαφάνεια, γιατί μειώθηκε στο 41%. Δεν το γνωρίζουμε. Άρα, μία από τι ε, προτάσει θα μπορούσε να είναι να προβαίνει σε μια ποιοτική αξιολόγηση ο διαμεσολαβητή στι περιπτώσει όπου αυτό είναι πιθανό. Και τέλο, η τελευταία σύσταση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ε, περιπτώσεων ε, στις οποίες ο διαμεσολαβητής ε, εμφανίζεται ενώπιον του Σολομέλεια στο Κοινοβουλίου. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και πια, κάποια πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα ζητήματα, για παράδειγμα το αν θέλουμε τελικά να μεταβάλουμε τη φύση του διαμεσολαβητή ή όχι. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο κάτι τέτοιο συνάδει με την προσπάθεια που κάνετε τώρα εδώ, αλλά για παράδειγμα μια δυνατότητα που έχει συζητηθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι να έχει τη δυνατότητα ο διαμεσολαβητής να παραπέμπει υποθέσει στο δικαστήριο. Και εδώ βέβαια κάτι τέτοιο έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ε, το πλεονέκτημα θα ήταν ότι οι αποφάσεις πλέον του διαμεσολαβητή θα έχουν άλλο βάρος, αλλά το μειονέκτημα θα ήταν ότι υπάρχει ο κίνδυνος όλες αυτές οι περιπτώσεις δηλαδή διαφοράς με ένα διοικητικό όργανο, με ένα θεσμικό όργανο να ε, οδηγούνται τελικά ε, σε, σε, δίκη, σε δικαστική διαδικασία. Και ε, όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς η αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή κινείται πέραν της ε, νομιμότητας, αν θέλετε, ε, ε, όπως αυτή καταγράφεται στις συνθήκες. Οπότε το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα μόνο να εξετάζει από νομική άποψη ζητήματα νομιμότητα. Οπότε, αν δίναμε μια τέτοια περισσότερη εξουσία στον διαμεσολαβητή, τότε βέβαια το δικαστήριο δεν θα μπορούσε να εξετάζει όλα αυτά τα ζητήματα της γκρίζα ζώνης που μπορεί σήμερα να εξετάζει ο διαμεσολαβητής. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.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 από την πλευρά του διαμεσολαβητού ε, ε, χρησιμοποιώντας και επί τη βάση των ήδη προβλεπομένων ε, στις συνθήκες και εν πάση περιπτώσει οι όποιες αλλαγές να μην γίνουν ξαφνικά αλλά να είναι βαθμιές και πιο μαλακές κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε πολύ καλά τα είπε ο κύριος Χαουρέγγι επίση και στα συμπεράσματά του. Αυτή η μεγαλύτερη εμπλοκή ας πούμε και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα ε, και όλα τα υπόλοιπα που είπε ο συνάδελφος με βρίσκουν απολύτως ε, σύμφωνοι. Και με τον τρόπο αυτό ε, θα έχει όλες τις εξουσίες που πρέπει, όλες τις αρμοδιότητες ε, που έχει και οπωσδήποτε την έγλη του, του λειτουργήματός του. Ε, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, όλες τις οδούς μπορούμε να τις ε, διερευνήσουμε. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο, Τζόρτζ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω κάποια ερωτήματα στην κυρία Κοτανίδη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Και με περιέργεια ε, άκουσα ε, να αναφέρεται ε, το θέμα των οργανισμών, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που με απασχολεί ήδη στα πλαίσια της δικιάς μου έκθεσης. Περιπτώσεις κακής διοίκησης υπάρχουν ή που να συνδέονται με τους οργανισμούς και πώς παρουσιάζονται. Δεύτερον, Είπατε beyond legality, πέρα από την νομιμότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτός ο όρος. Ε, αν, αν δεν περιλαμβάνει την ε, παρανομία ή την μη νομιμότητα, ε, τότε θα περιλαμβάνει κάποια γκρίζα ζώνη. Με εκπλήσει λίγο και με προβληματίζει αυτή, αυτός ο ορισμός. Αλλά ας πούμε και ότι τον δεχτώ αυτό το beyond legality. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να ξεπεράσει σε συγκεκριμένες διαδικασίες, να ξεπεράσει την τυπική νομιμότητα και κατά κάποιο τρόπο να ε, άρει αυτό το πέπλο έτσι ώστε να προσπαθήσει να βρει την ε, ίστατη αλήθεια, ας πούμε. Επίσης, υπάρχει ένα ε, σώμα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταγγέλλοντες εάν έχουν προβλήματα με τη διοίκηση. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ομπουτσμέν ε, των διαμεσολαβητών. Πώς λειτουργεί αυτό, Πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει, ας πούμε, μία ιδέα από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο επίπεδο των κρατών μελών ή αντίστοιχα, αντίστροφα. Υπάρχει κάποια, ας πούμε, λίστα βελτίστων πρακτικών. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, η διαδικασία ε, να είναι αμφίδρομη και επίσης υπάρχουν και διορθώστε με αν λαθεύω κάποια κράτη μέλη που δεν έχουν ε, διαμεσολαβητή. Θα τους αφήσουμε στην άκρη. Τι γίνεται τι γίνεται με την Γαλλία ή το σύστημα το οποίο από ό,τι θα ξέρετε φαντάζομαι ε, θα εγκατασταθεί ή θα δημιουργηθεί στην Ουγγαρία. Ε, επίσης το θέμα της αμέλειας. Νομίζω ότι δεν χρησιμοποιήσατε τον όρο αυτό με την νομική του υπόσταση και έννοια, αλλά με την έννοια της ε, κοινή λογικής. Δηλαδή κάτι που πρέπει να κάνει ένα συγκεκριμένο ε, όργανο και δεν το κάνει, ένας οργανός και δεν το κάνει, ή ας πούμε κάτι που πρέπει να ε, δοθεί ας πούμε στην, την πρώτη, να παραδοθεί την 1η Νοεμβρίου αλλά τελικά παραδίδεται την 17η Νοεμβρίου. Και αυτό μπορεί να ανήκει στις δικαιοδοσίες ας πούμε του διαμεσολαβητή. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Μία ερώτηση, κυρία Κοτανίδη. Κάπου στην Ευρώπη έχουμε ένα είδος μόνιμης ας πούμε επιτήρησης και reporting ε, όπως είχαμε ας πούμε για το κράτος δικαίου, για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Έχουμε κάτι που να μετράει ας πούμε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τον αριθμό των ε, υποθέσεων, έχουμε κανένα πίνακα επιδόσεων, scoreboard ή κάτι τέτοιο που να μας ε, δείχνει ε, την κατάσταση και τον ρόλο των εθνικών ε, διαμεσολαβητών. Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν, αφού έχετε όλες τις ερωτήσεις σε εσάς και μετά την Κομισιόν και πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε. In fact, the first question... Το πρώτο ερώτημα που είναι όμως ε, πολύ σχηδές, ελπίζω να θυμηθώ όλα τα στοιχεία του. Τα ε, ευρω... Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί βάσει των πληροφοριών που παίρνω από την ε, έκθεση του 16. Ο ίδιος ο διαμεσολαβητής λέει και αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του πόσες Ε, διαδικασίες ε, ε, the commission. Πόσες προσφυγές έχουν υποβληθεί σε σχέση με τους οργανισμούς. Επίσης βλέπουμε ακριβώς και τον τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι αφορά συλλογικά και ή τι αφορά κάθε μία, καθέναν από τους οργανισμούς την έννοια τώρα της κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, ε, πολύ γενικό ερώτημα. Εσείς ο ίδιος ε, είπατε τι υπάρχει πέρα από την νομιμότητα, beyond legality. Είναι γεγονός ότι θεωρούμε ότι ενεργεί η, ε, και, πράττει η διοίκηση, αλλά δεν είναι όλα ρυθμισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Μπορεί ε, να έχουμε την έννοια της ε, ελιπούς ή του ελιπούς εξυγχρονισμού της διοίκησης ή της, ε, της διοίκησης που δεν έχει εξυγχρονιστεί Αναφερόμαστε λοιπόν σε μία ε, διοίκηση η οποία θα είναι ανοιχτή, η οποία θα είναι συνεργατική και η οποία δεν θα πρέπει να δείχνει αμέλεια, δεν θα πρέπει να κρύβει ενδεχομένως κάποια έγγραφα και στα πλαίσια λοιπόν μιας σύγχρονης ε, διοίκησης ε, που δεν θα είναι περίκλειστη, ε, αυτά που λέμε έχουν έννοια. Αυτή είναι η ευρεία έννοια που δίνουμε εμείς στην κακή διοίκηση. Συνήθως έχουμε κάποια στοιχεία γραπτά ε, τα οποία συνηθίζουμε να τα έχουμε ε, ε, πολύ αυστηρά χωρισμένα. Αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό είναι άσπρο, αυτό είναι μαύρο. Αλλά πολλές φορές η κακοδιοίκηση μπορεί να είναι πολύ πιο λεπτή κατά κάποιο τρόπο και ο προσφεύγων μπορεί να ε, αναφερθεί σε κάποιον που δεν του έχει φερθεί ευγενικά ή που έχει αμελήσει κάποια από τα καθήκοντά του. Ναι, συμφωνώ πάντως μαζί σας ότι εδώ μιλάμε για μία γκριζόνη, αλλά ενδεχομένως αυτό είναι και το θετικό του υφισταμένου συστήματος, γιατί είναι γεγονός ότι μπορεί κανείς να βάλει σε αυτή την έννοια πάρα πολλά πράγματα, αλλά δίνεται και η δυνατότητα να αλλάξει το περιεχόμενο με τα χρόνια εάν ε, ε, μελετήσει κανείς ε, τη θητεία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου διαμεσολαβητή, βλέπουμε ότι έχει εξελιχθεί και το περιεχόμενο της κακοδιοίκησης. Ο πρώτος διαμεσολαβητής ήταν πολύ πιο δογματικός, ο δεύτερος πιο διευρυμένος και ο τρίτος πιο πολιτικός εντός εισαγωγικών. Κατά την έννοια αυτή δυσκολεύομαι να σας δώσω τελικό ορισμό, κλειστό ορισμό ε, της ε, κακοδιοίκησης και ο κύριος Ρανζέλ ε, πολύ σωστά τα λέει. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι και σίγουρη ότι απήντησα στην ερώτησή σας ή αν θέλετε ε, να σας πω και τίποτα άλλο. Είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στο Δινεκέ. Αν θέλετε να απαντήσετε στι υπόλοιπε ερωτήσει όμω. Εάν υπάρχει κάποιο φορέ που υπερισχύει, θα πρέπει κανείς να κοιτάξει τις αποφάσεις που προκύπτουν από το γραφείο του Δημοσιολαβητή. Από καιρού καιρών ε, συντάσσει κάποια έκθεση για, για την προσέγγιση που ακολουθεί ο διαμεσολαβητής σε υποθέσει. Αυτό προσδιορίζεται τρόπο τινά Ένας άλλος τρόπος μπορούμε να δούμε τη διαμεσολαβονομολογία που υπάρχει, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ε, μπορούμε απλώς να σκεφτούμε τις αιτήσεις εκθέσεις, που είναι αρκετά διαφωτιστικές. Ε, είναι σύντομη η εκδοχή που προκύπτει τα τελευταία χρόνια, συντομότερη από πριν. Μπορεί λοιπόν κανείς, διαβάζοντας τις εκθέσεις αυτές, να αντιληφθεί πώς αποφασίζει ο διαμεσολαβητής. Επίσης απαραίτητο είναι να θυμόμαστε ότι ο διαμεσολαβητής δεν επινοεί τίποτε. Απλώς τηρεί τον νόμο. Δηλαδή αποφαίνεται για την νομιμότητα. Δεν λειτουργεί εκτός νομικού πλαισίου ή θεσμικού πλαισίου. Εντός παραμένει και αποφασίζει αν ε, ακολουθήθηκαν, τηρήθηκαν οι αρχές. Και αν οι κανονισμοί και αρχέ αρχές της έγιναν σεβαστές αλλά και αν ακολουθήθηκε ας πούμε ο κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφορά. Για την άλλη σας ερώτηση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιολαβητών και Δημοσιολαβητριών. Το ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο ε, είναι αυτό που συνδέει το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς λειτουργεί. Λειτουργεί με έναν τρόπο ανεπίσημο δεν έχει στην πραγματικότητα θεμελιωθεί ως θεσμός. Λειτουργεί χαλαρά. Επικοινωνούμε μεταξύ τους οι δημοσιολαβητές. Πολλές φορές υπάρχουν κοινέ έρευνες, υποθέσεις που εξετάζονται από κοινού και αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον Η μελέτη βέβαια δεν στάθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας αυτού του δικτύου. Προς στιγμή είναι αυτά μπορώ να σας ε, παρουσιάσω. Ε, παραλήψεις, πλημελήματα, κακοδιαχείριση και ποια η σχέση μεταξύ τους. Ναι, η παράληψη κάποιας πληροφορίας. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με την διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε και πρέπει να τηρούνται. Και ο διαμεσολαβητή πάντοτε ελέγχει, εξακριβώνει κατά πόσο έγιναν σεβαστέ εξαιρέσει για την πρόσβαση στα εμπιστευτικά και απόρριτα έγγραφα και αν ακολουθήθηκαν σωστά οι κανόνε. Είναι λοιπόν κάτι που απασχολεί τον δημοσιολαβητή. Είναι υπάρχει ένα βαθμολόγιο ε, για τον δημοσιολαβητή, όπω είπατε, Πρόεδρε. Όχι εξ όσων γνωρίζω. Έχουμε λοιπόν ε, τις πληροφορίες αυτές και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για μερικά εκτός. Σας ευχαριστώ κύριε Κοτανίδας. Θα ήθελα να ζητήσω και από τον κύριο από τον υπεύθυνο του τμήματο για τα θέματα, τον μεσολαβητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα πει τη γνώμη του. Κοιτάξτε, είμαστε ο καλύτερο πελάτη του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή. 60% των υποθέσεων αφορούν εμά. Ε, να επιβεβαιώσω κάποια από τα πρακτικά πορίσματα τη έρευνα. Η τελευταία αριθμή που έχω από την Επιτροπή είναι ότι το 80% των υποθέσεων τη Επιτροπή τελικά δείχνουν ότι τηρούμε του κανόνε του Δημοσιολαβητή και 90, κατά 90% των υποθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή δείχνουν ότι κατά 90% ε, η τελική απόφαση του δημοσιολαβητή, το πορισμά του, δείχνει ότι δεν υπήρχε κακοδιαχείριση από πλευρά Επιτροπή. Γιατί κοιτάμε και το Λίνου, μέσα και τελευταία στιγμή. Μερικέ βέβαια υποθέσει έχουν προβληθεί πάρα πολύ στην κοινή γνώμη, γι' αυτό έχουμε κακό όνομα ε, και σίγουρα πετυχαίνει καλά αποτελέσματα ο Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή. Όμω στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε κάτι να το σκεφτούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ στο καταστατικό. Ακολουθούμε ως καλός πελάτης τη Μεσολαβητή τις συζητήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρητικά τουλάχιστον, και την όλη πολιτική συζήτηση για την ενδεχόμενη αλλαγή του καταστατικού. Όμως, εγώ εδώ δεν έχω εντολή να τοποθετηθώ για κανένα από αυτά τα σημεία. Βασική ανησυχία της Επιτροπής πάντως είναι όλα να παραμένουν εντός του θεσμικού πλαισίου όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ παυλου εχω Έχω δύο-τρεις τελευταίες παρατηρήσεις. Δεν θα σας εκπλήσει που θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτό που ο Γεώργη Σόπφιν. Είναι σαφές παρεπιπτόντος ότι ο Δημοσιολαβητής πέραν της νομιμότητας μπορεί να αξιολογήσει εάν τηρούνται αρχές καλής διαχείρισης, καλής διακυβέρνησης, συμπεριφοράς και διαγωγής των θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι κλασικό. Είναι κλασική αρχή του γερμανικού δικαίου. Ε, είναι κανόνε που υπάρχουν αυτοί, αλλά υπάρχει και αναλογικότητα και τρόπον την αυτό είναι νόμιμο. Είναι σαν ένας ε, συμβατικός γάμος. Ε, οπότε εδώ υπάρχει περιθώριο παρέμβαση του διαμεσολαβητή. Αλλά δεν μπορεί να αποφανθεί και για όλα. Για μένα αυτό είναι σαφές. Είναι η ουσία της έννοιας της κακοδιαχείρισης μάλιστα. Κατά δεύτερον, στον ε, συνάδελφο Χουαρέχη να πω ότι όντω βάσει κάποιων συστημάτων ε, ο διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και στο δικαστήριο. Μπορεί ο Πορτογάλος διαμεσολαβητής, ας πούμε, έχει το δικαίωμα να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, όπως είπατε, αυτό είναι απόρρια του παλιού συστήματος. Διότι στην Πορτογαλία, λόγω χάρη, στο Πορτογαλικό Σύνταγμα, δεν έχουμε τη Verfassungsbeschwerde, Οπότε ο διαμεσολαβητή μπορεί να λάβει ε, προσφυγές από του πολίτες και αν θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν παραδεκτές να τις πάει στο δικαστήριο. Δεν θα πάω τώρα στο αμερικανικό σύστημα που θα ήταν ίσως μια λύση για αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι στην περίπτωση του δικού μας συστήματος το καλύτερο είναι ο διαμεσολαβητής να μείνει εκτός δικαστικής αιθούσης. Αυτό πρέπει να το σκεφτώ περισσότερο βέβαια. Και για να ολοκληρώσω, Νομίζω ο Μοντεσκέ στις περσικές επιστολές του το 1779 νομίζω ήταν ε, έλεγε και τη φράση ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε κάτι με τρεμάμενο χέρι Νομίζω αυτό είναι ένας άγραφος κανόνας. Τι ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα κουμπάμε μόνο με τρεμάμενο χέρι, ακροθυγός τέλος πάντων. Ναι, να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης αυτής. Εξέταση στις 6 Δεκεμβρίου Πάουλου. Θα είσαι έτοιμος φαντάζομαι. Μετά προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών 13 και ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ 22 Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου περνάει στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να επαναλάβω, συνάδελφοι, κάτι που ίσως δεν έφτασε στα αυτιά σας ε, το πρωί κανονικά. Οπωσδήποτε τον Απρίλιο και τη δεύτερη του Μαρτίου θα έχουμε μόνον ψηφοφορίες θα είναι μπούκτη ολομέλεια για νομοθετικά θέματα. Μπορεί να ισχύσει και για την πρώτη του Μαρτίου. Όλες αυτές οι εκθέσεις που έχετε πάνω στα γραφεία σας και δεν έχουν νομοθετικό περιεχόμενο πρέπει να ολοκληρωθούν Γενάρη και Φλεβάρι. Οι δεν θα περάσουν καθόλου. Ε, κατανόηση λοιπόν παρακαλώ. Ε, τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Μετά περνάμε στα θέματα του Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Περνάμε στο 13 της ημερήσιας διάταξης. Αυτή τη φορά πρέπει εγώ να σας ενημερώσω που έχουμε πάει με το Brexit και τι είναι το κενό. Και να σας πω ότι δεν, εάν δεν συμβεί κάτι εξαιρετικά αρνητικό μέχρι την επόμενη συνάντηση, δηλαδή την επόμενη Τρίτη, θα έχουμε τη συνάντηση της ε, ΑΦΚΟ με το Task Force υπό τον ε, Πανιώτο ώστε να ακούσουμε μια λεπτομερή παρουσίαση των όσων ήδη γνωρίζουμε ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εξέβρεση μιας οριζόντιας συμφωνίας και την σχετική δήλωση. Την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή μετά από την προηγούμενη ενημέρωση που σας έκανα, στις 12 του μήνα, υπήρξε χθες μια συνάντηση και in camera με τα μέλη δηλαδή του Steering Group ε, και από εκεί και μετά και με τον Επίτροπο Μπαρνιέκε συζητήθηκε καταρχήν ε, βασική, τα βασικά μηνύματα αν θέλετε που περιλαμβάνονται μέσα στην πολιτική δήλωση και ακούστηκαν ένα σωρό από διαφορετικά σχόλια τα οποία υπόθηκαν από τις διάφορες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες ε, δεν έχουν κάποιους εκπροσώπους μέσα σε αυτήν την ομάδα καθοδήγησης το Steering Group. Εγώ αναφέρθηκα κυρίως στη σημασία τη μεγαλύτερη διαφάνεια που χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση αυτή τη διαδικασία και επίση αναφέρθηκα και στα κεφάλαια του level playing field, δηλαδή των ίσως, ίσων όρων του παιχνιδιού, αν θέλετε. Ε, επίση αναφέρθηκα στο ζήτημα τη. Ε, ε, της, ε, λήψη αποφάσεων με οριζόντιο χαρακτήρα και όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιότητα ε, τη δική μα Επιτροπή. Στη συνάντηση από εκεί και μετά με τον κύριο Μπαρνιέ, ε, υπογραμμίσαμε τη σημασία της παρουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και του ρόλου του σε ό,τι αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Μικτής Επιτροπής. Και αναφερθήκαμε και στο ζήτημα της σύνθεσης της Μικτής Ομάδας. καθώς αυτή θα είναι και αρμόδια, η κυρίως αρμόδια ομάδα για την παρακολούθηση της ε, ε, διαδικασίας εφαρμογής της συμφωνίας στην οποία θα έχουμε φτάσει και κατά συνέπεια ε, θέλουμε να υπάρχει και κατάλληλη εκπροσώπηση σε αυτή την ομάδα που του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αναφέραμε στον κύριο Μπανιέ. Επίσης αναφερθήκαμε και στο ζήτημα ε, της παράτασης της σχετικής προθεσμίας, δηλαδή ως προς το τι ακριβώς σημαίνει και πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, πάντοτε συμμορφούμενοι με τη συνθήκη. Επίσης συζητήσαμε κάποια ακόμα ζητήματα τα οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. αλλά τα οποία για παράδειγμα δεν, για τα οποία δεν έχουμε ενημερωθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή σε κάποια σημεία γνωρίζουμε περισσότερες ε, λεπτομέρειες ενώ σε κάποια άλλα δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες στη διάθεσή μας. Επίσης την τελευταία εβδομάδα βρέθηκα στο Κόζακ ε, στη Βιέννα, την Δευτέρα δηλαδή, όπου έκανα μια ε, διάρκεια σε ό,τι αφορά το Brexit και ήρθα σε επαφή και με συναδέλφους από τη, σε σχέση με το ε, Brexit και βρέθηκα ανάμεσα σε δύο πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές και οι αντιδράσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν πολύ θερμές σε ό,τι αφορά δηλαδή την, την στάση τους απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή υπήρξε, εκφράστηκε λύπη για αυτή την ε, αποχώρηση αλλά και σεβασμός. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις διμερείς συναντήσεις είχαμε με συνάντηση ε, με την Ένωση των Μικρών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι και ιδιαίτερα σημαντική γιατί βέβαια ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, έχουν προβεί σε κάθε είδους σχεδιασμούς έκτακτης ανάγκης για τον Brexit, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά δηλαδή την δυνητική αποχώρηση από την ενιαία αγορά, από την Τελωνιακή Ένωση και ούτω καθεξής, γιατί βέβαια θα χάσουν ως τρίτη χώρα την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, ήρθα, ε, συναντήθηκα και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον ε, Τουρισμό και τον Πολιτισμό του Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου και το οποίο συζήτησε και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον Brexit. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι πριν από μία εβδομάδα ολοκληρώσαμε, οριστικοποίησαμε ε, την συμφωνία αποχώρησης και από εκεί και μετά έγιναν κάποιες συζητήσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο και όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση υιοθέτησε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε αυτή την ε, πολύ ε, δύσκολη συζήτηση που έγινε στην Κάτω Βουλή με την Πρωθυπουργό Μέη και από εκεί και μετά βέβαια η βασική περίληψη της ε, πολιτικής ε, δήλωσης και η ίδια η συμφωνία ε, δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά οπότε έχουν υφίσταται στην ιστοσελίδα ταυτόχρονα διανεμήθηκαν και σε όλα τα μέλη της μέλη της ΑΦΚΟ και βέβαια η συμφωνία αποχώρησης είναι 135 σελίδες ε, αλλά το outline, δηλαδή η περίληψη, είναι μόνο 20 σελίδες. Ε. Από εκεί και μετά, ε, στην διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη, συναντηθήκαμε και πάλι με το Steering Group για τον κύριο Μπαρνιέρ και έγινε ακριβώς αυτή η συζήτηση σε ό,τι αφορά την συμφωνία αποχώρησης. Και επίσης θα ήθελα να σας καλό να ρίξετε μια ματιά στην Συμφωνία Αποχώρησης, ώστε να μου πείτε τι ακριβώς ε, χρειάζεστε να μάθετε περαιτέρω, δηλαδή σε ποια σημεία χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, γνωρίζετε πως υπάρχουν έξι τμήματα στην Συμφωνία αποχώρηση, κάποια από τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας, για κάποιου από εμά. Εδώ αναφέρομαι για παράδειγμα στο, ιδιαίτερα στο ζήτημα των δικαιωμάτων των ε, πολιτών ε, και βέβαια το ζήτημα της τη. της του οικονομικού του διακανονισμού, πράγμα το οποίο θεωρούσαμε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα τελικά στο οποίο καταφέραμε να ε, φτάσουμε σε μια συμφωνία σχετικά γρήγορα. Και μετά βέβαια το ζήτημα των ε, γεωγραφικών ενδείξεων και το ε, ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, τα ζητήματα στα οποία καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία όπως βέβαια και το ζήτημα των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αλλά ε, και βέβαια έχει τεθεί το ζήτημα της ε, ενδιάμεσης ε, προθεσμίας το οποίο έχει προσελκύσει πολύ ενδιαφέρον και βέβαια έχει αποτελέσει την πηγή παρανοήσεων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως η μεταβατική περίοδος το ενδεχόμενο της οποίας είχε επιτρέψει από την αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθύ εξ αρχή, ε, υπό ορισμένε προποθέσει, ε, τελικά δείχνει να αξιοποιείται από την ε, Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτό ακριβώς για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο νομικό κενό που θα μπορούσε να προκύψει ανάμεσα στην ημερομηνία αποχώρησης του, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη Τη ισχύω της νέας συμφωνίας που θα διαδεχτεί, δηλαδή που θα ρυθμίζει το νέο καθεστώς. Άρα λοιπόν καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά αυτή την προθεσμία παράταση, για την οποία επίση συμφωνήθηκε ότι θα μπορούσε να παραταθεί περαιτέρω, άπαξ και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και βέβαια θα πρέπει εδώ να πληρούνται συγκεκριμένε προποθέσει. Ότι δηλαδή ε, το δυναμικό, αν θέλετε, υλοποίηση τη νέα συμφωνία ε, θα είναι ήδη ορατό στον ορίζοντα και με βάση αυτή την, ακριβώς αυτό το εφικτό τη νέα συμφωνία θα χορηγηθεί η νέα παράταση. Ε, και βέβαια εδώ δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα αν θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη περίοδο, αν θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά αυτό νομίζω πως θα εξαρτηθεί από τη Βρετανική κυβέρνηση σε σχέση με το τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω πως η κυρία Μέη μεταβαίνει προς τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Γιούνκερ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί και η πολιτική δήλωση. Όπως ακούσαμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ε, η, η έκτακτη διάσκεψη κορυφή τη Κυριακή έχει προβλεφθεί όχι για πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά για την επίσημη, αν θέλετε, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση τη διαδικασία. Ε, γιατί να θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Οπότε να δούμε μέχρι τότε τι θα έχει επιτυχθεί. Πάντω η πολιτική δήλωση είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για μα, αλλά και για τη Βρετανική πλευρά και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας στη Βρετανική πλευρά. Αλλά ε, αναλαμβάνω ότι η πολιτική δήλωση δεν είναι ε, νομικό κείμενο, αλλά πραγματικά πολιτικής φύσης έγγραφο. Θα έχουμε λοιπόν στη διάσκεψη κορυφή την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων και από εκεί και μετά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά την κύρωση. Δηλαδή, από την Βρετανική πλευρά υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να τρέξει και την γνωρίζουν καλύτερα οι Βρετανοί συνάδελφοι, αλλά για μα εδώ, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το επωνομαζόμενο Meanful vote. Ε, αυτή η ψηφοφορία λοιπόν επί της ουσίας και όσο το ταχύτερο λάβει αυτή η χώρα τόσο ε, ταχύτερα θα μπορέσουμε να κινήσουμε και τη δική μας διαδικασία. Και ποια θα είναι αυτή θα πρέπει να λάβουμε τη σχετική αναφορά από το Συμβούλιο, το οποίο δηλαδή θα απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο με το αίτημα της έγκρισης της συμφωνίας αυτής, δηλαδή έγκριση, δεν ξέρω πώς το ακριβώς το, το, ορμάζει συνθήκη, και θα κληθούμε να δώσουμε είτε καταφατική είτε αρνητική απάντηση, ναι ή όχι. για το ίδιο θα ισχύσει και για το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και μετά από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμφωνία πηγαίνει και πάλι στο Συμβούλιο καθώς εμείς θα χρειαστούμε απλή πλειοψηφία εδώ για να εγκρίνουμε, ενώ στο επίπεδο του Συμβουλίου θα ε, υπάρξει ειδική πλειοψηφία. Θα προσπαθήσει να κινηθεί βέβαια προς την ομοφωνία, αλλά δεν θα είναι απαραίτητη η ομοφωνία. Και βέβαια η διαδικασία στη Βρετανική πλευρά είναι περίπλοκη και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα πριν από τα τέλη Μαρτίου. Αυτά λοιπόν μπορώ να σας κοινοποιήσω σήμερα, αυτά γνωρίζω. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια καλή εβδομάδα. Αλλά όταν κοιτάω το Ρίτσερτ, Ε, πραγματικά δεν μπορώ να αναφέρω τη λέξη επιτυχία σε ό,τι αφορά δηλαδή, την επιτυχή έκβαση ε, των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία, γνωρίζοντα ότι αυτή η συμφωνία αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά ε, σίγουρα είναι καλό το ότι, να, ε, ότι έχουμε μια συμφωνία, γιατί πραγματικά η μη ύπαρξη συμφωνία δεν είναι αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι θα υπάρξει δηλαδή κάποια άλλη έμεση οποία συμφωνία. Όχι, πραγματικά θα είναι απουσία συμφωνία σε ό,τι αφορά δικαιώματα πολιτών, σε ό,τι αφορά όλα τα ε, ζητήματα. Και από εκεί και μετά η ύπαρξη μια συμφωνία δημιουργεί και μια ε, ένα θετικό κλίμα, ένα κλίμα εμπιστοσύνη θετικό σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Γιατί φαντάζομαι ότι και κλεισμένο των θυρών κάποιοι δηλαδή ήδη εργάζονται επί της ε, μελλοντικής εντολής ε, και το τι θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Απριλίου. Εν πάση περιπτώσει πότε ακριβώς ελήγει τότε 29 Μαρτίου η προθεσμία. Οπότε ε, παρότι πρόκειται για, μια, ε, για το Brexit, το οποίο δηλαδή ε, δεν είναι προ όφελο ούτε τη μία πλευρά ούτε τη άλλη, ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε μια θετική συμφωνία. Ο συνάδελφο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω μόνο το εξής, γνωρίζοντας ότι ε, εξαρτώμεθα και από την διάσκεψη κορυφή ε, της Κυριακή και βεβαίω κυρίω και από την πολιτική δήλωση που θα ακολουθήσει τη συμφωνία. Δεν ξέρω εάν οι συνεδρίε που έχουμε προβλέψει για την επόμενη εβδομάδα μήπως λέω, θα ήταν ενδιαφέρον για την Επιτροπή μα ΑΦΚΟ να έχει την δυνατότητα να συζητήσει με έναν εκπρόσωπο των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω εάν αυτό το έχει ήδη αναφέρει. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Ε, είπαμε, είπα στην αρχή, ότι εάν δεν συμβεί κάτι περίεργο και αρνητικό και απρόσμενο, τότε θα, έρθουν στη, θα έρθει ε, κάποια, θα έρθουν κάποια μέλη τέλο πάντων τη διαπραγματευτική ομάδα του κυρίου Μπαρνιέ την Τρίτη. Α, ναι, εγώ νόμιζα ότι θα κάναμε συνεργασία με την ε, Steering Committee. Α, ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία τότε. Special, right. Mm-hmm. Ε, Where's Madame James? Oh, he's over there. Yes, please, Diane James. Κύριε Diane James. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος ε, βέβαια της ε, Brexit Committee ε, και δεν μου επέτρεψαν να συμμετάσχω και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε ο κ. Μπαρνιέ. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι παράπλευρο. Νομίζω ότι το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη πόσο άσχημα υποδέχτηκε το, η Μεγάλη Βρετανία το, η συμφωνία, αυτό το deal και δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά όταν ακούει κανείς ε, την ομάδα του Μπαρνιέ ε, να φουσκώνει σαν το Γάλλο και σαν τη Γαλοπούλα και να, ε, ειδικά ένας Γερμανός από την ομάδα του να αναρωτιέμαι ίσως κάποιος που είναι στην steering committee Ίσως θα πρέπει να το μεταφέρει αυτό το σχόλιο, δηλαδή να δούμε τι γίνεται και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Επανέρχομαι πάντως ε, ότι γίνεται ε, μεγάλη επίκριση, πολλές επικρίσεις ακούμε από την συμφωνία. Ναι, βεβαίως ακούω και το αντεπιχείρημα ότι δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε, να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο, το κατανοώ και αυτό. Αλλά τις τελευταίες 48 ώρες ε, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ε, προσπάθεια δυναμήτησης αυτής της συμφωνίας με τον κύριο Μπαρνιέ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ας πούμε, ε, ξεπέρασε τα δικά του εσκαμένα και είπε ότι η Σκοτία θα μπορούσε να μείνει ή να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση των όσων έχουν συμφωνηθεί. Δεύτερον, με μεμονωμένα ε, μέλη τα οποία θέλουν να ε, αφαιρέσουν πλήρως την Συμφωνία Αλίας και αυτό γιατί θέλουν πρόσβαση στα είδατα της, Ευρωπαϊκής, της ε, Μεγάλης και τρίτον το γεγονός ότι πλέον έχει προκύψει, έχει εγερθεί ζήτημα για το Γιβραλτάρ ε, και σε σχέση με ενδεχόμενες ε, εμπορικές συμφωνίες. Επομένως, όσοι λένε ότι πάρα πολύ ωραία είναι όλα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως θα πρέπει να τους πω ότι να το ξαναδούνε λίγο. βεβαίως να συγχαρώ την γραμματεία του ΑΦΚΟ γιατί έκαναν ένα έγγραφο πάρα πολύ ε, ενδελεχές ε, έγγραφο και το λέω σαν ε, θετικό. Γιατί από την Βρετανική πλευρά δεν είχαμε ούτε μισή πληροφορία. Ε, σίγουρα ίσως στους φιλοευρωπαίους να έδωσαν κάποια ψυχία, αλλά οπωσδήποτε όχι στους ευρωσκεπτικιστές. Ναι, ξέρετε, λέει η Πρόεδρος, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν περαιτέρω στο μέλλον. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συζητήσεις. Ε, είπατε και στην αρχή Ε, ε, ε, ότι στην αρχή όντως υπάρχει με σημαντικές περιπτώσεις πολύ μεγάλος υπερβολικός θα λέγαμε ενθουσιασμός και αυτό είναι να αποφεύγεται. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε δει αντίστοιχε κινήσεις και αντίστοιχε ελεκτικές υπερβολές και από τους Brexiteers όταν ε, ε, χτυπούν την κυρία Μέι, Μέη, Νομίζω ότι ε, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα αν ε, δεν είχαμε και deal, γιατί θα βρισκόμαστε σε ένα είδος ε, χώρου limbo και δεν θα, θα υπήρχε κανένα, καμία βάση συζήτησης σε σχέση με τα όσα ε, λαμβάνουν χώρα και το διάλογο στη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία, η Πρωθυπουργό λέει είτε θα πάρετε τη δικιά μου συμφωνία είτε ε, επέρχεται καταστροφή. Γι' αυτό έχουν προκληθεί και τόσες πολλές ε, αντιδράσεις. Είναι λίγο στο στυλ το δέχεστε ή αλλιώς καταστραφόμαστε ή αυτό ή τίποτα. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο αυτή η δυτή ε, ε, επιλογή ε, και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι πρόκειται για μια κακή συμφωνία. Υπάρχουν οι ευρωσκεφτικιστές οι οποίοι ενδεχομένως οποιαδήποτε συμφωνία θα την θεωρούσαν αρνητική και οτιδήποτε μπορεί ακόμα να του συνδέει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι de facto κακή συμφωνία. Ωστόσο είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι είναι κακή η συμφωνία όσον αφορά ας πούμε τη δήλωση για το μελλοντικό πλαίσιο όσο έχει τώρα είναι στην ουσία μας οδηγεί σε ένα τυφλό Brexit, δηλαδή φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Και επιμέρους διαφετιστικές συζητήσεις ε, μεταφέρονται για ύστερη, μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Δεύτερον, βγαίνουμε από την ε, Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διατάξεις για προσωρινή ε, παραμονή στην ε, Τελωνιακή Ένωση, που όμως είναι σαφές ότι είναι πρόσκαιρη και για όσο γίνεται μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε και θα υπέρθει η απόσυρση από την ε, Συμφωνία, την Τελωνιακή Ένωση, συγγνώμη. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα σαφές σύνορο ε, και επομένως απειλείται η ε, ε, απρόσκοπτη ροή εμπορευμάτων από τη μία πλευρά των συνόρων στην άλλη. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε με, ένα, με ελέγχου στα σύνορα, με ένα σκληρό σύνορο, με δασμούς, νέες επιβολές δασμών και ειδικών φόρων κτλ αποτέλεσμα όλων αυτών των διάφορων σημείων και των επικρίσεων δεν είναι πολύ πιθανό να εγκρίνει η Βουλή ε, τον Δεκέμβριο τη συμφωνία αυτή. Και με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει κρίση. Κρίση βεβαίως στην Βρετανική πολιτική σκηνή κρίση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί ναι, φαντάζομαι ότι η ευρωπαϊκή πλευρά ε, θα περιμένει απλώς να δει τι θα γίνει, αλλά θα περιμένει με αδημονία και με αγωνία και με άγχος. Ε, υπάρχει βέβαια και το βασικό αφήγημα ότι για όλα αυτά είναι οι Βρυξέλλες και αρκεί κανείς ε, να ρίξει το φταίξιμο στις Βρυξέλλες για να τη βγάλει καθαρή, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να δούμε τι κάνει και η, Ευρωπα... τι κάνει, ε, και η Βρετανική κυβέρνηση και τι έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ίσως δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν το θέμα λόγω δικών τους εσωτερικών διαφορών. Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν καθαρά. Εάν απορριφθεί λοιπόν αυτή η συμφωνία, εξακολουθεί να παρεμένει μια τεράστια πλειοψηφία ε, στο, στη Βρετανία που δεν θέλει να αποσυρθεί η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τη στιγμή που θα έχει προκύψει μια συμφωνία και θα έχει αποσυρθεί, τι μέλη γενέστε. Ε, η μία οδός θα ήταν ε, επαναδιαπραγμάτευση διαφορετικής συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βέβαια προς ώρας ότι όχι, όχι, εμείς δεν ανοίγουμε καμία νέα διαδικασία και καμία νέα διαπραγμάτευση. Αλλά ίσως να υπάρχει κάποια λογική προσφορά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πλευρά ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και τότε ίσως τα πράγματα να αλλάξουν. Υπάρχει λοιπόν μία συμφωνία που δεν είναι αποδεκτή, υπάρχει όμως και η αρχή ότι ε, δεν μπορεί, ε, ε, ότι, δεν μπορεί να φύγει κανείς χωρίς μία συμφωνία και επομένως και επομένως θα πρέπει κάπως να ξαναδούμε τα πράγματα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν θέλουν ε, να φύγει η Βρετανία. 700.000 ε, ε, διαδήλωσαν στο Λονδίνο πρόσφατα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ ευμετάβληπτη η κατάσταση. Και αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτήν την μεταβλητότητα και αυτό το ευμετάβληπτο της ε, ε, κατάστασης. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς και άλλοι είπαν ότι σέβεστε την απόφαση ε, που μέσω του δημοψηφίσματος πήρε ο Βρετανικός λαός. Άρα, ακριβώς εμείς ως δημοκράτες σεβόμαστε την επιθυμία ε, του λαού, θα πρέπει να σεβαστούμε και οποιαδήποτε έκφραση μεταβλημένης γνώμης έχουν ε, οι Βρετανοί. Δηλαδή, αν έχουν αλλάξει άποψη, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η άποψη αυτή, η τροποποιημένη. Σας εξέθεσα λοιπόν τις απόψεις μου, αλλά και μία ερώτηση. Η Steering Group ε, τι, για τον Brexit προτίθεται να εγκρίνει ψήφισμα τον ε, Δεκέμβριο μετά από το, τη διάσκεψη του Δεκεμβρίου. Όχι, δεν νομίζω για, την, για το Δεκέμβριο για τη διάσκεψη Ορυφή. Δεν ξέρουμε. Εξαρτάται από το πώς θα πάνε τα πράγματα και πότε θα τον αναλάβει ΑΦΚΟ. Γιατί για την αναπομπή δεν ξέρουμε τίποτα. Θα πράξουμε αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Για την ώρα δεν υπάρχει απόφαση. Σπινέλη. Μετά την παρέμβαση του συναδέλφου ήθελα να πω ότι είχαμε, πήγε στην Κόζακ, Ντανούτα. Μίλησες με Ισπανούς βουλευτές και μεγάλους πρώτα για το θέμα του Γιβραλτάρ και μετά για το θέμα της αλίας που αφορά τους Γάλλους. Εξέφρασαν καμιά άποψη. Ε, εντόπισαν κάποια έλλειψη για την ώρα στη συμφωνία, ιδιαίτερα για το Κεβραλτάρ και την Αλία. Όχι. Κανείς. Δεν ανέφερε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μάλιστα η συμφωνία Αλίας, που είναι σημαντική για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για την πρόσβαση στα χωρικά ύδατα, αλλά και για την πρόσβαση στις αγορές, είναι κοινά τα συμφέροντα και θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Όπως ξέρετε, η μεταβατική συμφωνία θα είναι το status quo εκτό από τη συμμετοχή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων στα θεσμικά όργανα. Θα έχουμε το, τη δυνατότητα να το συζητήσουμε το μέλλον τη Ελία, είναι μέρο του μέλλοντο η Αλία. Για το Γιβραλτάρ ελπίζω να επιτευχθεί συμφωνία, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη, στην εξέβρεση λύση εκτό από ένα θέμα που δεν έχει λυθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει επιλογή. Λύση πρέπει να βρεθεί. Οι διαπραγματεύσει είναι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανία. Συνεχίζονται εδώ και μήνε και ελπίζω ότι είμαστε κοντά στην εξέβρεση λύση. Αλλά κανεί δεν έχει θέσει το θέμα. Πρέπει να πω ότι η εντύπωσή μου ήταν ότι τα εθνικά κοινοβούλια στις ομιλίες τους τοποθετήθηκαν περισσότερο πολιτικός ε, για τις δεσμεύσεις τους, για την πολιτική διάσταση όχι απλώς εκφράζοντας ε, την ε, δυσαρέσκειά τους ή τη θλίψη τους, αλλά ε, περισσότερο εκφράζοντας και την δική τους σχέση με την Βρετανική πλευρά. Δεν υπήρχαν τόσες λεπτομέρειες και είναι και φυσιολογικό αυτό, διότι τα Εθνικά Κοινοβουλία δεν έχουν ρόλο στην ε, υποστήριξη αυτή τη συμφωνίας δεν συμμετέχουν. Θα συμμετάσχουν σε μια δεύτερη φάση, στη μελλοντική συμφωνία. Θα είναι συμφωνία με τρίτη χώρα, τις χώρες μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε εκεί νομίζω θα υπάρξει μεγαλύτερη δραστηριότητα και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, πολλές συζητήσεις και συνεννοήσει κυβερνήσεων και εθνικών βουλών. Για την ώρα είχα την εντύπωση ότι δεν ήταν πολλά τα κράτη-μέλη που είχαν φοβερή γνώση του όλου θέματο. Την όλη τη διαδικασία τη προετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι για την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα ή που δεν θα υπάρξει συμφωνία. Γιατί και αυτό, αυτό ακόμη και για μένα είναι κάτι που με εκπλήσει. Ενώ έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοχεύουμε να επιτευχθεί συμφωνία βέβαια, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Ο Πασκάλ Αρντίνη, διευθυντής από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, νομίζω τον Ιούλιο, μίλησε για την όλη διαδικασία της ε, ετοιμότητας, πώς συντονίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ενημέρωσε και την περασμένη εβδομάδα μόλις εξηγώντα όλες τις λεπτομέρειες του θέματος της ετοιμότητας. Έχω πάντως την εντύπωση ότι δεν είναι ένα ζήτημα που είναι ευρέως γνωστό σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. κυρία Ντότζ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν εδώ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας ε, από την αρχή. Ήταν μια φοβερά φορτωμένη περίοδος στο γραφείο μου, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε για αυτό το θέμα που εγείρει τόσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα, να συζητιέται με τρόπο γεμάτο σεβασμό σε αυτό το διάλογο μεταξύ συναδέλφων και ίσως και με αποχρώσεις κάπως διαφορετικές από τον τόνο που είχε η όλη συζήτηση στη δική μου περιοχή του Ηνωμένου Βασίλειου και γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Πρόεδρε, ωστόσο, ζούμε σε καιρούς περίεργους. Εγώ ήρθα εδώ, στην Επιτροπή αυτή σήμερα, στη συνεδρίασή μας, και πραγματικά βρίσκομαι ε, σε φάση και δεν το λέω με καμία διάθεση να προκαλέσω να συμφωνώ με τον κύριο Κόρμπετ. Δεν είναι καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να φτάνουμε να το πούμε αυτό από πολύ διαφορετικέ σκοπιέ, Ρίτσαρτ, αλλά πραγματικά δεν είναι καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίση συμφωνούμε ότι ο Πρωθυπουργό, έτσι όπως έχει περιγράψει τη συμφωνία και θέτει στους ανθρώπους την επιλογή ναι ή όχι, άσπρο ή μαύρο, είναι ψευδοεπιλογή, ψευδοδήλημα. Η Πρωθυπουργό μας λέει ή η συμφωνία μου ή το χάος. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διπλή επιλογή είναι λανθασμένη και μπορούμε να την ε, βελτιώσουμε αυτή τη συμφωνία και να τη διορθώσουμε. Και όπως φαντάζεστε, θέλω πολύ συγκεκριμένα να μιλήσω για τη Βόρεια Ιρλανδία και για τη συμφωνία Backstop. Στην ε, Βόρεια Ιρλανδία πολλοί κόσμοι έρχεται και μου λέει γιατί επικεντρώνεστε διαρκώ στο μηχανισμό Backstop διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι ε, η ουσία των μελλοντικών μας σχέσεων. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε γιατί εκεί θα καταλήξουν. Και μου λένε μη κάθεστε και σκάτε για τον backstop, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε ακριβώς έτσι. Ο μηχανισμός του backstop θα ισχύει για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ως τελωνιακός διακανονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και κάποιο σχολιαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι ο... η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι στο βάθος του τούνελ αυτού του διακανονισμού και το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ε, στο πάνω μέρος ε, της ε, πλευράς αυτή, του καναλιού αυτού. Και κάποιος άλλος είπε ότι ο τελωνιακός κώδικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμένει ευθυγραμμισμένη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την νομοθεσία για τα ΦΠΑ, τους ειδικούς πόρους κατανάλωσης και συγκεκριμένα αγαθά. Θα ισχύουν οι ίδιοι υγειονομικοί κανόνες για τη γεωργική παραγωγή, για την θέση σε εμπορία και για τις κρατικές επιδοτήσεις. Αλλά αν δούμε την συμφωνία την ίδια και το πρωτόκολλο, από τη δική μου την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, 68 σελίδε αφιερώνονται στην περιγραφή αυτών των κανόνων. Ε, Κανόνε, του οποίου θα πρέπει να προσυπογράψει η Βόρεια Ιρλανδία και που θα μα κάνει να διαφέρουμε από τα άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό και πάλι, τι περίεργη κυρία, όπω είπε και ο Τζέρεμι Κόρμπιν ε, σήμερα. Ε, τι περίεργο να δημιουργείται αυτό το νοητό σύνορο στην Ιρλανδική, στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Η Βόρεια Ιρλανδία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι σχεδόν τρίτη χώρα από την άποψη της νομοθεσίας. Οπότε αρχίζει κανείς να αντιλαμβάνεται γιατί το κόμμα μου θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι καλή ούτε για τη Βόρεια Ιρλανδία ούτε για την συνοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ως κράτους. θα ξεπηδήσουν ένα σωρό προβλήματα για την Βόρεια Ιρλανδία. Η Ηνωμένη, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη αγορά για μα. Πουλάμε περισσότερα εκεί από ότι στον υπόλοιπο κόσμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και στη δημοκρατία τη Ιρλανδία μαζί. Είναι η αγορά από την οποία αγοράζουμε τα περισσότερα αγαθά μα. Και με μια αυξανόμενη απόκληση με τον καιρό θα είναι δύσκολο να γίνει κανονική πρόσβαση στην εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είμαι από αυτούς που συμφωνούν με την ιδέα ότι θα ήταν ίσως καλό ε, να αφήσουμε να εκτελεχθεί ένα, μια πιθανότητα, ένα σενάριο ε, καμιάς συμφωνίας, μηδενικής συμφωνίας ε, στα παρασκήνια. Το κόμμα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι και οικονομικά σταθερό και όλη μας περιοχή το ίδιο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλουμε καμία συμφωνία ή να ξεφύγουμε. Θέλουμε τη σωστή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τη Βόρεια Ιρλανδία. Και για τους γειτονέ μου ε, από την άλλη πλευρά της θάλασσας της Ιρλανδίας και τους γειτονέ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, εμείς δεν την υποστηρίζουμε αυτή τη συμφωνία γιατί δεν είναι η σωστή. Ευχαριστούμε κυρία Ντότς, ο κύριος Χουαρέγγι. Ήθελα να ξεκαθαρίσω στην κυρία Ζέμφια και στην Μπάρμπαρα Σπινέλη το εξή αυτά που έλεγαν χώρα ε, από πλευρά τη Ισπανική κυβέρνηση σε σχέση με αυτή την πιθανή συμφωνία. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε μονάχα διευκρίνηση όσον αφορά το περιεχόμενο συγκεκριμένου άρθρου σε σχέση και με μία αρχή η οποία είχε γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί στις ε, guidelines της διαπραγμάτευσης που είχαν γίνει δεκτές ε, ήταν ξεκαθαρισμένο ότι το μελλοντικό καθεστώς του Γιβραλτάρ σε σχέση με την Ευρώπη θα ε, έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση απευθεία ανάμεσα στην στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία άποψή μας είναι ότι ενδεχομένως αυτή η αποσαφήνιση, η διευκρίνηση χωρίς κανένα πρόβλημα ε, θα ενσωματωθεί στις δηλώσεις και επομένως δεν θα υπάρχει πρόβλημα και από τη μεριά ε, της Ισπανίας. Ευχαριστούμε πολύ ο Γιολάιενεν. Ναι, νομίζω πως καθίσατε σαφές πως υπάρχουν ακόμα μία σειρά από προβληματικά σημεία και αδιέξοδα. Πάντως, ε, για μένα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πριν από εβδομάδες ακουγόταν ήδη, 5-6 εβδομάδες, ότι σε τεχνικό επίπεδο είχαμε καταλήξει ήδη σε συμφωνία. Δηλαδή, ήδη οι εμπειρογνώμονες είχαν καταλήξει ως προς το τι ακριβώς είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Και είχαν λοιπόν συμφωνήσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, αυτός ο διαχωρισμός, ο συνοριακός δηλαδή, της Βόρειας Ιλανδίας με την Ιλανδία και επίσης δεν μπορεί να υπάρξει cherry picking, δηλαδή επιλογή των στοιχείων που θα θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά. Δηλαδή, όταν βγαίνει από την ε, ενιαία αγορά, είναι εκτό ενιαίας αγοράς Ωστόσο, δείχνει με αυτή την άποψη των εμπειρογνωμών να μη συμφωνεί ε, ο κόσμος της πολιτικής γιατί φαίνεται πως υπήρξαν και κάποιε ψευδεστήσει, αλλά και δεν υπήρχε και επίγνωση του ποια θα ήταν τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν με τον Brexit. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον της πραγματικότητας. Ότι δηλαδή θέλουμε να σεβαστούμε την ε, συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Άρα θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη λύση και από την άλλη αυτό που αναφέρεται ότι θέλει κανείς να βγει από, τον, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ταυτόχρονα θέλει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ε, και αυτή είναι η δεύτερη, αν θέλετε, ψευδέστηση που υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να είναι εκτός και ταυτόχρονα να είναι εν μέρη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ε, πως αυτό που λένε ε, και ο Κόρμπιτ βέβαια είναι σωστό. Δηλαδή ότι ε, δεν είναι ικανοποιητικό αυτό το αποτέλεσμα. Και εγώ θα το έλεγα αυτό, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με Brexit χειρότερο είναι από την τωρινή κατάσταση. Οπότε σε κάθε περίπτωση δηλαδή με τέτοια συμφωνία δεν είναι ικανοποιητική. Εντάξει, ο Ρίτσαρντ βέβαια ε, έχουν διαφορετικό σκεπτικό, δηλαδή ο Ρίτσαρντ και η Γεραντότση, ωστόσο το συμπέρασμα είναι το ίδιο, ότι η συμφωνία δεν είναι ικανοποιητική. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το blind Brexit, ένα σκληρό δηλαδή τυφλό Brexit και το κατά πόσο χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο. Ε, ναι, στα τέλη Μαρτίου θα λάβει χώρα η έξοδο, αν δεν λάβει κάτι άλλο χώρα μέχρι τότε. Και από εκεί και μετά θα χρειαστούμε περαιτέρω χρόνο σε ό,τι αφορά την σύναψη μια νέα συμφωνία. Αλλά εάν σε μια τέτοια διαδικασία θέλουμε να συμμετάσχουν όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα 27 εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, τότε προφανώς θα χρειαστούμε τον απαραίτητο ε, χρόνο. Θα χρειαστεί λοιπόν παράταση της μεταβατικής περίοδου. Και πολλά μπορούν να συμβούν. Πολλοί δηλαδή, πολλά πράγματα έχουν να συμβούν ακόμα, μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Άρα λοιπόν, Αυτά τα δύο στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω. Ότι από τη μία πλευρά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να έχουμε μια ικανοποιητική συμφωνία γιατί το Brexit από μόνο του αυτό καθεαυτό αποτελεί επιδείνωση σε σύγκριση με την σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ. Al de los comentarios de la... Δεν είχα σκοπό να παρέμβω, αλλά άκουσα αυτά που, μου, που είπε η κυρία James και νομίζω ότι ε, καλό είναι να γίνει μια διευκρίνηση. Να τα δούμε ένα-ένα. Συμφωνούμε ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα ε, και εκείνη αναφέρεται σε μεγάλα προβλήματα από πλευράς ε, κρατών, κρατών μελών, αλλά αυτά είναι ελάσσονο σημασίας. Αναφέρθηκε άλλωστε και πριν. Το ε, κύριο πρόβλημα είναι ότι θα περάσει στην ιστορία των διαπραγματεύσεων ότι η διαπραγμάτευση ενός απέναντι σε 27 έχει 27 ενωμένους με ε, συνένεση, ενώ από την πλευρά του ενός γίνεται το έλα να δεις. Δεν ξέρω να το πω διαφορετικά. Menos daño a nuestra... Και ε, εμείς ε, με τις διαφορές μας, τις οικονομίες μας, ε, στα δικαιώματα κτλ. Καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι. Εάν όμως η Βρετανική πλευρά δεν είναι ενωμένη, δεν έχει δηλαδή έναν μύτο αριάδνης από την αρχή μέχρι το τέλος της διαπραγματεύσεις, μα τότε δεν γίνεται να επιτύχει κάτι η πολιτική, η κοινωνία, ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε το δημοψήφισμα που δεν είχε έτσι καλά ε, καθορισμένες αρχές, που δεν είχε καλά καθορισμένες ε, πλειοψηφίες και ειδικέ πλειοψηφίες κλπ. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν θα είναι η ενωσιακή πλευρά, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτή που θα έχει αποτύχει, γιατί εμείς ξεπεράσαμε πολλά βάζοντας πάνω απ' όλα το κοινό συμφέρον και με όλο το σεβασμό σας λέω ότι σας τα λέω όλα αυτά. Εγώ θέλω να ολοκληρωθεί η συμφωνία όσο γίνεται πιο καλά. Αλλά πραγματικά θα καταγραφεί στην ιστορία των διαπραγματεύσεων ότι είχες έναν από τη μία και 27 από την άλλη, ο ένας διαλυμένος με τον εαυτό του και οι 27 ενωμένοι όλοι. Και το λέω πραγματικά από τα βάση της καρδιάς μου με μεγάλη αγάπη. Σας ε, ο κύριος Σέφλιν. Το είπα και προηγουμένως, αλλά νομίζω αξίζει να το επαναλάβω. Έχει κρίση συνταγματικού χαρακτήρα το Ηνωμένο Βασίλειο. νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι οργανωμένο έτσι. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε πόσο απρόσμενη είναι όλη η διαδικασία που έχουμε ζήσει από το δημοψήφισμα και μετά. Και επίσης να πω και το εξή. Τρίτα κράτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, όποια και αν είναι η έκβαση αυτή τη συνταγματική κρίση, θα είναι ένα πολύ διαφορετικό τρίτο κράτο από το οποιοδήποτε άλλο. Όχι μόνο για λόγου παραδοσιακού ιστορικού και γειτονία, αλλά γιατί έχει υπάρξει κράτο μέλο δημιουργείται ένα διαφορετικό σκηνικό. Θα πρέπει να συλλογιστούμε τι θα πει αυτό το καθεστώς τρίτου κράτους. Θα φανεί με το χρόνο βεβαίως, αυτό είναι προφανές, αλλά πρέπει να το σκεφτεί η επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Και αυτό θα με φέρει στο επόμενο σημείο μου, που μπορεί να σας φανεί κάπως επιπόλαιο. Μετά τις 29 Μαρτίου, θα είναι αρμοδιότητα της ΑΦΚΟ το Brexit. Θα το δουν οι Ίντα και Άφετ, ε, υποψιάζομαι, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να μην το χάσουμε κι εμείς. Άντερσον. Είναι ενθαρρυντικό που ξέρει το Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι πραγματικά σημαντικό η διαπάλη μεταξύ διαφορετικών ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τέλος πάντων, πέρα από τα χιούμορ. Όταν έχει κανεί πολιτική εξουσία και έχει την πλειοψηφία και κυβερνάει, εάν του συμβεί κάτι κακό, τι θα σκεφτεί ο κόσμος, ότι φταίει. Δεν έχει καμιά σημασία αν είναι όντως το δικό, δική του η ευθύνη ή όχι. Ο κόσμος θα σκεφτεί, εσείς έχετε την εξουσία να προσέχατε, να τα πάτε καλύτερα, για να αποφευχθεί αυτό το στραβό που έγινε. Μπορεί να πει κανείς ότι η μερίδα του λέοντος ε, της ευθύνης για την ενδεχόμενη και εγώ ακόμη θέλω να πιστεύω ότι είναι ενδεχόμενη η περίπτωση και υπόθεση να υπάρξει μηδενική συμφωνία. Σίγουρα ε, είναι ευθύνη λοιπόν της ΜΕΗ και του, πάρτι, του κόμματος των Τόριδων. Μιλάμε για ένα σενάριο που θα έχουμε δύο πλευρές και δεν είμαι βέβαιος ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοβούλια ε, θα ε, έχουν προσπαθήσει να διευκολύνουν την κυρία Μέη. έχει πολλά προβλήματα και αυτή την κακή παρτίδα τη χειρίστηκε και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ένα Brexit που να είναι ένα τροχαίο, σαν ένα σοβαρό τροχαίο. Δηλαδή μην φτάσουμε να καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Είναι και σενάριο υψηλού κινδύνου. Η οικονομική καταστροφή μπορεί να μας χτυπήσει και θέλουμε να την αναχαιτήσουμε. Πρέπει όμω να είμαστε και προετοιμασμένοι να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε, Μάρξ. Μπάρμπαρα Σπινέλη, τελευταία στον κατάλογό μου. Συμφωνώ μάλλον με αυτά που είπε η Diane Ντόντς. Είναι περίεργη κύριε. Δίκιο έχετε. Ωστόσο, αυτό που είναι παράδοξο είναι ότι είναι περίεργη και ταυτόχρονα πολύ ορθολογιστική. Είναι πλούσιοι και παράξενοι όπως την καταιγίδα του Σέξπιρ. Γιατί λέω ότι είναι και ορθολογιστική και πλούσιοι. Διότι για το μηχανισμό backstop της Βόρειας Ιρλανδίας η συμφωνία απόσυρσης πρέπει οπωσδήποτε να είναι, ε, σε, να με άλλες διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες και, όλες, και πιο συγκεκριμένα τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Εάν δεν είναι συνεπής, θα έχετε πάλι την απειλή του πολέμου και σοβαρότατες εντάσεις μεταξύ Αγγλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. ή θα γίνει δημοψήφισμα στη Βόρεια Ιρλανδία για να επανενωθείτε με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αυτό θα ήταν θετική έκβαση. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτά τα προβλήματα της ε, συνέπειας με τις διεθνείς συνθήκες. Εάν εγκριθεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και αυτό θα είναι το πρόβλημα για τη δική σας πολιτική δύναμη. Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσω με αυτό που ο Μαξ Άντερσον. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποφύγουμε το σοβαρό τροχαίο. Διότι αν υπάρχουν τόσες ε, αντιστάσεις στη συμφωνία από εσείς, τότε είναι αλήθεια, και ρωτώ τους φίλους από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για την απουσία συμφωνίας στην Αγγλική Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι αλήθεια. Πείτε μου. Ευχαριστώ. Πασκάλ Ντιρό. Πασκάλ Όχι. Α, ου. Ντανούτα, ούτε και εγώ δεν ήθελα αρχικά να πάρω το λόγο, αλλά δεν θέλω ε, να ακουστεί μονάχα αυτού του είδους ε, η, ε, αυτού του είδους το σκεπτικό από τη μεριά των πρασίνων, δηλαδή ότι δεν βοήθησε το Κοινοβούλιο την Τερέζα Μέη. Δεν είναι σωστό να λέγεται αυτό, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, αλλά και ιδιαίτερα ο Μισελ Μπαρνιέ, αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών έκαναν τα πάντα για να προσπαθήσουν να επιτύχουν έχουμε να επιτευχθεί μια ε, συμφωνία εποφελής και για τις δύο πλευρές, ένα deal καλό και για τους δύο. Και είναι εκπληκτικό που δεν έχουμε εδώ το θάρρος να αναφέρουμε ότι ε, ότι η πολιτική τάξη, ε, υπήρχε μια πολιτική τάξη ολόκληρη στο Ηνωμένο Βασίλειο που είπε ψέματα στους πολίτες τους, είπε ε, αν βγούμε θα γίνει αυτό ή το άλλο. Πολλοί Βρετανοί στην ακρόαση μας είχαν πει ότι ιδίω στην Ιρλανδία θα εφευρίσκεται ένα σύνορο 2,0 και ρωτήσαμε τότε, μα τι είναι αυτό το σύνορο 2,0 εγώ δε, επίσης δεν καταλαβαίνω, ίσως είμαι ένας απλοϊκός Γάλλος, αλλά ποτέ δεν μου εξήγησαν και ούτε το κατάλαβα, ούτε ποτέ στη φυσική, ούτε στη λογική, ούτε στα μαθηματικά να είναι κανείς και μέσα και έξω. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι κάποιος είπε ψέματα στον ε, Βρετανικό λαό. Και τώρα ερχόμαστε να ε, ε, πούμε ε, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και ότι κάποια στιγμή εμείς γίναμε υπεύθυνοι, κατέστημεν υπεύθυνοι για την κακή κατάσταση και όχι αυτοί με τις εθνικιστικές τους κορώνες. Ε, εμείς θέλουμε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τίποτε άλλο. Εγώ πραγματικά δεν είμαι θρησκευόμενος. Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα. Δεν πιστεύω στο δυσυπόστατο ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι και μέσα και έξω και εδώ και εκεί. Εγώ ξέρω ότι ε, υπάρχουν άνθρωποι στην ε, Μεγάλη Βρετανία, στην κυβέρνηση της κυρίας Τερέζα Μέη, που την ε, κρατούν όμοιρο και συγγνώμη για την βαριά αυτή έκφραση. Ε, και πραγματικά το γεγονός ότι έχουν αλλοπρόσαλη και αμφιλεγόμενη διαρκώς ε, και αλληλοανερούμενη στάση από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι δικό μας ε, σφάλμα και δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Δεν δέχομαι και δεν δέχομαι και ούτε σαν κοινοβούλιο αλλά και σαν ομάδα των Πρασίνων να αφορέσουμε αυτό το καπέλο και αυτή την ευθύνη. Ευχαριστώ. Κυρία Ντότς. Κυρία Ντότς και μετά να τελειώσουμε. Thank you um, for allowing me to come back. Σας ευχαριστώ που μου αφήνετε να ξαναπάρω το λόγο και θα είμαι πολύ σύντομη. Πάντως, νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Ε, αναφερθήκατε στο ότι η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να συνάδει με άλλες διεθνείς συμφωνίες και φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στη συμφωνία του Μπέλφαστ ή στη συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής όπω είναι γνωστή δηλαδή ευρύτερα η συμφωνία του Μπέλφαστ. Ακριβώ λόγω τη ημέρα που υπογράφηκε. Και αναφέρατε επίση ότι τα ζητήματα ε, των συνόρων θα πρέπει να επιληθούν με ένα συνεχτικό τρόπο. Αν διαβάσετε αυτή τη συμφωνία του Μπέλφαστ δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το ζήτημα των συνόρων. Δεν είναι δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται στην ελόγω συμφωνία. Και από εκεί και μετά ένα άλλο επιχείρημα το οποίο ακούω επανειλημμένα από διαφόρου είναι ότι το ότι αν θέλουμε ε, ε, να αποφύγουμε ένα σκληρό σύνορο, όπως είπαμε, αυτό το hard border. Ε, και εγώ πραγματικά ε, βρίσκομαι 15 λεπτά από τα σύνορα. Δηλαδή, αν μπω στο αυτοκίνητό μου και οδηγήσω σε 15 λεπτά, θα έχω διαβεί τα σύνορα. Και για μένα, λοιπόν, είναι πραγματικά συμφέρον, αποτελεί συμφέρον μου το να μην υπάρξει αυτό το hard border, το σκληρό σύνορο. Όμως, αυτό το σκληρό σύνορο υπήρξε στο παρελθόν και υπήρξε προκειμένου ακριβώ να ε, προβούμε σε πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές. Άρα νομίζω πως δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε τα σύνορα του παρελθόντος με τα σύνορα ε, που έχουμε σήμερα, δηλαδή ένα σύνορο τελωνιακό και ένα σύνορο αγαθών. Και από ό,τι γνωρίζω πρόκειται για ένα οικονομικό ε, σύνορο, ένα σύνορο ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα νομισματικό σύνορο. Από τη μία πλευρά έχουμε ευρώ, από την άλλη πλευρά έχουμε στερλίνα και αγγλική λίρα. Και σε προηγούμενη παρέμβαση είχα αναφέρει ότι υπάρχουν σελίδες επί σελίδων με διατάξεις που θα ισχύσουν για την ε, Βόρειο Ιρλανδία, αλλά δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολιτικός ηθήνων ο οποίος θα μπορέσει είτε να συμφωνήσει είτε να διαφωνήσει με τις εν λόγω διατάξεις όπως αυτές θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποια ήταν η βασική αρχή που, η οποία χαρακτήριζε ακριβώς τη Συμφωνία του Belfast αυτή η, δυνατότητα της συνένεση των δύο κοινοτήτων, δηλαδή το να μπορούν να συνενέσουν οι δύο κοινότητες αυτό που συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία η οποία παραγνωρίζει ε, την παράγραφο 50 ε, του κειμένου το οποίο συμφωνήθηκε από κοινού ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την, από την Βρετανική κυβέρνηση ουσιαστικά ακριβώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή παραγνωρίζεται ε, αυτή η βασική αρχή της συνένεσης που αποτέλεσε τη, βασική αρχή της συμφωνίας του Belfast. Ε, και να σας πω εγώ από την πλευρά μου ότι εγώ ότι δεν ψήφισα υπέρ τη συμφωνία του Μπελφαστή, τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Και έχω εξηγήσει επανειλημμένα το γιατί. Γιατί ε, βγήκαν άνθρωποι από τη φυλακή οι οποίοι είχαν προβεί σε τρομοκρατικέ ενέργειε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν βομβαρδίσει, άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκοτώσει. Και εγώ δεν ήμουν σε θέση λοιπόν να συμφωνήσω, να υπερψηφίσω μια τέτοια συμφωνία. Και δεν μπορούσα να προτείνω κάτι τέτοιο στους ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν εμένα ως πολιτική εκπρόσωπο σε σχέση με αυτήν την συμφωνία. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, πολύ σύντομα και εσείς, παρακαλώ. Πολύ σύντομα να πω ότι οι προσπάθειες που κάνει η Βρετανική πλευρά για να πει ότι εκείνο που φταίει, ότι το φταίξιμο βρίσκεται στην πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εντελώ εσφαλμένο. Εκείνο που φταίει, τουλάχιστον κατά 99%, είναι η Βρετανική κυβέρνηση. Άρα, όπω κάνετε, εγώ συμφωνούμε κατά 99,9%. Αλλά εάν συμβεί κάτι άσχημο, Και εδώ τώρα δεν παίρνω το λόγο εκ μέρου των ε, Πρασίνων, έτσι. Παίρνω το λόγο ω Ευρωβουλευτή, αλλά μέλο των ε, Πρασίνων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι το αρνητικό. Ελπίζουμε να έρθει στα λογικά της η Βρετανική κυβέρνηση, αλλά ε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ε, δώσαμε το λόγο σε όλου του συναδέλφου που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή, αλλά βέβαια δεν θα έχουμε εξαντλήσει όλα αυτά τα ε, ζητήματα που θα θίξετε και την επόμενη εβδομάδα. Ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μα και η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή ΑΦΚΟ θα λάβει χώρα 27 Νοεμβρίου. Θα είναι ολοήμερη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ.